Bene colleghi, possiamo cominciare? I ε, συνάδελφοι, παρακαλώ να ξεκινήσουμε. Σας παρακαλώ καθίστε, γιατί έχουμε, έχουμε πολλές υποφορίες. ανακοινώσεις. Καταρχήν έγκριση μάλλον της ημερήσιας διάταξη. Αν συμφωνείτε, ωραία, το εγκρίνουμε. Έχουμε διερμηνία από πολλέ και διάφορες γλώσσες. Και ευχαριστώ εκ των προτέρων του διερμηνείς. Και να σας πω ότι αναμεταδίδεται στο ίντερνετ η συνεδρίασή μας και επίσης σας καλώ να συμμετέχετε στις 6 Μαΐου στο μεσημεριανό διάλειμμα στο σεμινάριο της ΤΟΑ για το πώς η τεχνολογία θα μπορούσε να αλλάξει τον τρόπο να διδάσκει κανείς και να μαθαίνει. Και αυτό συνδυάζεται με το δικό μας εργαστήριο που έχουμε προγραμματίσει για τις 4 Μαρτίου μαζί με την DG Connect και την DG ε, Εκπαίδευση που ακριβώς αφορά την ε, εκπαίδευση και την κατάρτιση στο ψηφιακή εποχή. Ε, επίσης, να σας ευχαριστήσω για τη στήριξη που δώσατε στην προφορική ερώτηση για το θέμα της καταστροφής του πολιτιστικού, ε, της πολιτιστικής κληρονομιάς στο Ιράκ και θα ήθελα η ομάδα σας ε, να στηρίξουν και το αίτημα που έχω ήδη υποβάλει, ώστε η απάντηση στην προφορική ερώτηση να ε, γίνει στην επόμενη σύνοδο του Στρασβούργου, γιατί θεωρώ ότι είναι επίγον. Τώρα, να παρακαλέσω επίσης όλες τις ομάδες. Τι γίνεται, υπάρχει κάποιο πρόβλημα μετάφρασης? Όχι. Λοιπόν, η Επιτροπή, ε, της Επιτροπή, του Πολιτισμού και οι ομάδες σας να στηρίξουν τις θετικές ε, εμπειρίες, με πλήρη βέβαια ε, διαφάνεια. Έγινε μια ψηφοφορία την Επιτροπή Κοντ που θέτει σε κίνδυνο το βραβείο Λούξ. Και θέλω εκεί να μας στηρίξετε. Ας προχωρήσουμε ε, ένα μικρό σύντομο ε, διορθωτικό για τα πολιτιστικά αντικείμενα ε, στις 26 Μαρτίου σας έγραψε η Γραμματεία προτείνοντας, ε, παρουσιάζοντας μάλλον ε, το σχέδιο τροποποίησης για το άρθρο 17 της Οδηγίας για την επιστροφή των πολιτιστικών αγαθών που ήδη έχουμε συζητήσει και εκεί έχει προσθεθεί μόνο η φράση κείμενο σχετικό με το κείμενο σχετικό με το και είναι μόνο μία ε, τροποποίηση. Αν δεν υπάρχει πρόβλημα, πρόβλημα το εγκρίνουμε άμεσα και θα, θα περάσει από την επόμενη ολομέλεια και εντό των επόμενων 24 ωρών θα τη θεωρήσω ότι εγκρίνεται αυτή η αλλαγή εάν δεν υπάρξουν αντιρρήσεις. Σας ευχαριστώ για την κατανόησή σας και θα περάσουμε αμέσως στις ψηφοφορίες όπου έχουμε τρεις σημαντικές ψηφοφορίες. Η πρώτη είναι της έκθεσης της Σιλβί Γκυγιώμα, την οποία ευχαριστώ για την εργασία της, σχετικά με την εξαιρετικά <clears throat> σημαντική, το σημαντικό θέμα του τροποποίησης του κανονισμού 1304-2013 όσον αφορά την αύξηση του ποσού της αρχικής χρηματοδότησης το οποίο καταβάλλεται στα επιχειρησιακά προγράμματα που στηρίζονται από την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων. Eh, να δώσω το λόγο στην εισηγήτρια καταρχήν πριν αρχίσουμε την ψηφοφορία και θυμίζοντα το εξή. Είδα ότι έγινε δεκτό το αίτημα τη εισηγήτρια να αποσυρθούν οι τροπολογίε ώστε να εγκριθεί αμέσω σήμερα ε, η έγκριση στην ΕΜΠΛ. Δηλαδή, ελπίζουμε ότι στην επόμενη συνεδρίαση την ε, διακόπτη Πρόεδρος, η κυρία Γιγιώμα, ευχαριστώ Σίλβια, είπες ε, τα βασικά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στο αίτημά μου να αποσύρουν τροπολογίες. Εγώ συμμερίζομαι απόλυτα την εργασία που έγινε. Θα σας ευχαριστήσω για τη συλλογική εργασία που έγινε. Απλώς θα ήθελα να πω το εξής. Ζήτησα από πολλές τις ομάδες να ανταποκριθούν στο αίτημά μας για το δήλωση που ζήτησα να κάνω. Οι πάντες πλην ενός ανταποκρίθηκαν. Σας ευχαριστώ και μπορούμε τώρα να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία. Έχετε όλοι τα τους καταλόγους ψηφοφορίας και ξεκινάμε. Τροπολογία 1. Με συγχωρείτε. Ναι, όχι, λέω το αντίθετο. Ναι, ε, ε, είπαμε ότι δεν έχει τροπολογίες. Λοιπόν, άμεσα η ψηφοφορία για το σχέδιο χνομοδότησης ε, ολόκληρο με, ηλεκτρονική ψηφοφορία άρχεται η ψηφοφορία. Ποιοι είναι υπέρ, ποιοι είναι κατά, ποιοι απέχουν να ψηφίσουν. Chiudo la <laughs> <laughs> Τέλο Τέλος της ψηφοφορίας. Πολύ ωραία. Έχουμε τα αποτελέσματα. Καλό αποτέλεσμα είναι γιατί έχουμε 24 υπέρ, μία αποχή και κανέναν κατά. Οπότε εξαιρετική η έγκριση που θα περάσει και από την Επιτροπή ΕΜΠΛ <clears throat> σήμερα. Περνάμε στη δεύτερη έκθεση στη συναδέλφου Ιζαμπέλα Αντινόλφη για την οδηγία του 2001 για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του, του copyright δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων. Έχετε εδώ αντιρρήσεις, όχι. Λοιπόν, περνάμε στη ψηφοφορία άμεσα και έχουμε τροπολογίες. Έχουμε την τροπολογία 1. Καταρχήν, ποιος είναι υπέρ.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 13 υπέρ, 14 κατά, απορρίπτεται. Τροπολογία 6. Υπέρ. Όχι, 7, γιατί η 6 έχει καταπέσει. Ωραία. 7 λοιπόν, τροπολογία 7. Κατά αποχές απορρίπτεται. 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 9 υπέρ αποχές νομίζω πως απορρίπτεται αλλά θα το ελέγξω ε, ηλεκτρονική ψηφοφορία λοιπόν για την 9 άρχεται Πάλι είναι ένας υπεράριθμος στο ΕΛΚ παρακαλώ. Αφαιρέστε μία κάρτα. Εντάξει τώρα. Τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Περνάμε στο 10. Ε, Υπέρ. Υπέρ κατά Έλεγχος. Απορρίπτεται με 17 ψήφους κατά. Τροπολογία 11. Ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 12 της εισηγήτριας υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 13 και 14 που είναι ταυτόσιμες υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 15 υπέρ κατά συγγνώμη πρέπει να πάμε στη 17 γιατί ε, αυτές έχουν ε, αυτή έχει καταπέσει λοιπόν 17 είναι μια τροπολογία με προφορική τροπολογία οπότε εάν την εγκρίνουμε την εγκρίνουμε τροποποιημένη Είμαι κατά της προφορικής τροπολογίας, παρακαλώ. Control A questo Τότε αλλάζει και η ένδειξη ψήφου, γιατί για μένα που είμαι εισηγήτρια καθίσταται αρνητική. Μια ένδειξη. Ωραία, λοιπόν, το σημειώνουμε. Ψηφίζουμε την τροπολογία 17 χωρίς την προφορική τροποποίηση. Ποιοι είστε υπέρ, κατά, ηλεκτρονικός έλεγχος. Ψηφίσετε παρακαλώ. Τέλος ψηφοφορίας. Ε, passo quindi 19. Chi è Περνάμε στο 19. Στην τροπολογία 19 υπέρ κατά αποχές. Σας παρακαλώ σηκώνετε τα χέρια. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 20. Εντάξει, έλεγχος. Chiudo la votazione. Spero di Τέλος της Εγκρίθηκε. Είχε εγκριθεί. Τροπολογία 20. Ποιοι είναι υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. 21. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 22. Υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Πάμε στην 24 του εισηγητή. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, έλεγχος. Γιατί δεν είναι πολύ σαφές. Chiudo la votazione. Τέλος της ψηφοφορίας. Allora, 21 eh, a favore, <laughs> scusate, allora, 21 a favore, 8 contro. Εγκρίνεται. Ναι, ε, συμβαίνουν αυτά. Περνάμε στη συμβιβαστική 1. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 28 υπέρ. Κατά. Α, αποχές εγκρίνεται. 29 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 30 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 31 με προφορική τροπολογία υπαριθμών 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 32 που έχει τροποποιηθεί από την προφορική τροπολογία. 2. Α, είναι ταυτόσημες. Ωραία λοιπόν. Συμβιβαστική 2. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Α, τώρα η 39, συγγνώμη. Υπέρ, κατά, ε, αποχές ε, εγκρίνεται. Είναι ταυτόσιμο με τη 40, 41. Α, όχι, συγγνώμη, πάμε στην 42. Κράσνοντεύσκη. Υπέρ 42, τροπολογία 42, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 43 υπέρ κατά αποχές Νομίζω ότι απορρίπτεται και περνάμε σε ηλεκτρονικό έλεγχο. Άρχεται η ψηφοφορία. Chiudo la votazione. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται για μια ψήφο. Σαραντα που είναι ταυτόσιμα με την 50 και την 51 και την 52. 49, 50, 51, 52. 4 τροπολογίες καλύπτονται. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. 55 τώρα. Έλεγχο θέλετε για τη 49. Εντάξει. Ε, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Ναι, ήταν σαφέ. Λοιπόν, φτάνουμε έτσι στην 55, ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ, κατά, από εγκρίνεται, συμβιβαστική 4, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, πάμε στην 64, στην επόμενη σελίδα, 64 υπέρ, κατά, Αποχές απορρίπτεται 65 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 66 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται όχι, έλεγχος Άρχεται η ψηφοφορία Τέλος ψηφοφορίας Απορρίπτεται 67, συγγνώμη της εισηγήτριας υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 68 υπέρ κατά αποχές έλεγχος. Τέλος ψηφοφορία, ε, άρχεται η ψηφοφορία, συγγνώμη. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με μία ψήφο διαφορά. 69 πέρα κατά αποχές. Νομίζω πως απορρίπτεται, αλλά θα ελέγξω. Με συγχωρείτε, αλλά θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Πάντα ίσα ίσα στο τσίμα, τσίμα γίνεται η ψηφοφορία απορρίπτεται 70 υπέρ ποιοι είναι κατά αποχές έλεγχος πάλι ηλεκτρονικός άρχεται η ψηφοφορία τέλος της ψηφοφορίας 15 υπέρ. Εγκρίνεται. Πάμε στην 72. είστε είστε υπέρ, κατά, αποχές, έλεγχος. Νομίζω πάλι πως και εκεί είναι ίσα ίσα. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Με μία ψήφο διαφορά. Δεν είναι πολύ εύκολο αυτό. 74 της εισηγητρίας. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι υπέρ. Όχι. Τι έχει γίνει λάθος. Έκανα λάθος. Όχι, το ψηφίσαμε την 72. Ελέγξαμε την 72. Την 74 τις εισηγήτριες ψηφίσουμε τώρα. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 75 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία, τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 86. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Έλεγχος. Για την 86 ψηφίζουμε. 86 τέλος ψηφορίας απορρίπτεται. Εβδομήντα Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 79. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Α, με συγχωρείτε. Απορρίπτεται. Όντως. Ε, για να το κάνουμε άλλη μια φορά. Υπέρ. Ξανά, για την ίδια. Ε, κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ναι, απορρίπτεται. 80 της εισηγήτριας. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 81 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 73 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 7 στην επόμενη σελίδα συμβιβαστική 7 στην επόμενη σελίδα ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται περνάμε στην 90 Τροπολογία 90 που είναι ταυτόσιμη με την 91 και με την 92. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται. 90... Ε, όχι. Συμβιβαστική 8. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Έλεγχος. Έλεγχος ηλεκτρονικός. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Οπότε πάμε στην 98. Υπέρ ποιοι είναι, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 99 και 100 είναι ταυτόσιμες υπέρ, αποχές εγκρίνεται. 101 υπέρ, κατά, αποχές 102 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 103 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 104 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 105 υπέρ, κατά, έλεγχος. Ελέγχουμε για την 105. Τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται με μία ψηφοδιαφορά. Τώρα, 106 υπέρ. Κατά αποχές έλεγχος τέλος της ψηφοφορίας Κοιτάξτε, δεν σηκώνετε τα χέρια σας. Το λέω και στην από εδώ ομάδα. Λοιπόν, 107 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται, 108, όχι είναι ταυτόσιμη, συγγνώμη, 109, υπέρ, κατά, αποχές, Νομίζω πως εγκρίνεται, αλλά για να είμαστε σίγουροι, ελέγχουμε. Εγκρίνεται. Και περνάμε στην 113. Τρούπελ. Υπέρ. <clears throat> Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 100. Α, συγγνώμη. Ο συνάδελφος Μόργανο. Στην 114 Έχω ένα θέμα σε σχέση με το τι ισχύει στις νομοθεσίες. Εκεί όπου λέει μόνο από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές να αντικατασταθεί από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. Εγώ προσωπικά νομίζω πως μπορεί να γίνει δεκτό, γιατί έτσι αναφέρεται στις διάφορες ε, δομές που υπάρχουν στα διάφορα κράτη-μέλη. Εάν συμφωνείτε με αυτή την προφορική ε, τροπολογία, να ψηφίσουμε για την 14 πώς τροποποιήθηκε. Α, όχι, όχι, διαφωνείτε. Οπότε πρέπει να ψηφίσουμε την 114 χωρίς την ε, τροπολογία. Υπέρ λοιπόν ποιοι είναι. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. 115. Υπέρ. <clears throat> Κατά αποχές εγκρίνεται. 116. Υπέρ. Α, συγγνώμη, είναι ταυτόσιμη. 118. Συγγνώμη, το 116 είναι ταυτόσιμο με την επόμενη, όχι με την προηγούμενη, με την 117. Άρα τις ψηφίζουμε από κοινό υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. 118 ε, τις εισηγήτριες υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 119 ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 120 είναι ταυτόσιμη και πάμε στην 121. Υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία για το σχέδιο γνωμοδότησης ε, ε, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Ρεστίντα con 14 voti Απορρίπτεται με 14 ψήφους ε, έναντι 12 για 4 αποχές. Quindi non è adottata la... Απορρίπτεται λοιπόν η έκθεση, αυτό πολύ με στενοχωρεί. Μάλλον θα ήταν καλύτερο, ε, το ξέρω πως κάνατε τέτοια δουλειά κυρία Συγγήτρια, για συντονισμό, περισσότερη ίσως εργασία για συμβιβαστικές και σημεία ε, συνένεση είναι ευαίσθητο το κόσμο, συνειδητοποιώ τις δυσκολίες, αλλά και προσωπικά εκφράζω την, ε, την αλληλεγγύη μου με την ε, ηθικήτρια Αντινόλφη. Παρακαλώ, κυρία Αντινόλφη. Διοργάνωσα πολλές ε, συνεδριάσεις των σκιωδών ακριβώς για να μπορέσω να ευνοήσω τη συζήτηση, οπότε ε, νομίζω ότι έκανα ό,τι ήταν δυνατόν και απαραίτητο. Μάλιστα κατηγορήθηκα ότι ακολούθησα λάθο κανόνες για τη διοργάνωση ε, των συνεδριάσεων των σκιωδών εισηγητών, πράγμα το οποίο δεν είναι αλήθεια, δεν, δεν θα το ξανασυζητήσουμε λοιπόν, δεν κρατάω καμιά πικρία. Ευχαριστώ. Και εμένα με στεναχωρεί γιατί η Επιτροπή Πολιτισμού δεν θα δώσει κοινή γνωμοδότηση για ένα θέμα τόσο πολύ ευαίσθητο. Ε, θα πρέπει αυτό να μας προβληματίσει και για το μέλλον όταν πρόκειται για τόσο ευαίσθητα ζητήματα. Χρειάζεται αμοιβαία κατανόηση και να προσπαθήσουμε να βρούμε συνενέσεις. Είμαι βεβαία πως έγινε η προσπάθεια, ωστόσο είναι ένα θέμα όπου ίσως οι ευαισθησίες σε αυτή την Επιτροπή μα είναι ιδιαίτερε σε σχέση με το δικαιώματα του δημιουργού και τα συγγενικά δικαιώματα. Εν πάση περιπτώσει καταγράφουμε αυτό το αποτέλεσμα και περνάμε στην επόμενη ε, ψηφοφορία που αφορά Σε αυτή τη φάση, επειδή δεν μπορεί να λείπει η γνωμοδότησή μας ή οι γνωμοδοτήσεις μας από τις επιτροπές, η Επιτροπή Τζούρι, δηλαδή της κυρίας Ρέντα. Σας καλούμε να υποβάλλετε τις τροπολογίες σας να τις στείλετε στην Επιτροπή εκείνη, ώστε να μπορέσουμε να εκφραστούμε. Φαντάζομαι πως πολλοί από εσάς θα το πράξετε γιατί νομίζω πως είναι σημαντικό να υπάρξουν κάποια μηνύματα που θα προέλθουν από τη δική μας Επιτροπή. Σας ευχαριστώ και περνάμε στην έκθεση της συναδέλφου Τρούπελ. Όπως γνωρίζετε είναι ένα σημείο πολύ σημαντικό Πρόκειται για τι συστάσει σχετικά με τι διαπραγματεύσει για τη διατλαντική εταιρική σχέση εμπορίου και επενδύσεων. Ζητήσαμε πολύ συγκεκριμένε κατευθύνσει ώστε να γίνει σεβαστή η εξαίρεση πολιτιστική και όπω έχει γίνει και σε προηγούμενε ε, τέτοιε ε, συνεδριάσει. Ευχαριστώ πολύ την Χέλγα Τρούπελ για την εργασία της. Έχουν γίνει αρκετές τροπολογίες. Η προθεσμία ήταν η 9η Μαρτίου. Σας δίνω το λόγο, αν θέλετε να πείτε δύο λόγια. Ευχαριστώ. Και πάλι να υπογραμμίσω ότι κοινό μας συμφέρον είναι οι οπτικοακουστικές υπηρεσίες on και offline, τεχνολογικά ουδέτερες, ε, πρέπει να συντηρούνται, να ρυθμίζονται από τα κράτη-μέλη και αυτό είναι νομική δέσμευση ότι οι, οπτικο, ε, οι οπτικοακουστικές υπηρεσίες δεν καλύπτονται από την ε, συμφωνία TTIP. Επίσης θέλουμε η συμφωνία αυτή να αναφέρεται στην δυνατότητα σταθερών τιμών για βιβλία ή και περιοδικά και νομίζω ότι είναι σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε ότι το TTIP δεν πρέπει να επηρεάσει τη δυνατότητα των κρατών μελών να υποστηρίζουν και να ρυθμίζουν θέματα εκπαίδευσης με ε, κρατική χρηματοδότηση ή με άλλη μορφή. Και αν υπάρχουν ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, αυτά θα πρέπει να πληρούν τα ίδια ε, κριτήρια ε, διαπίστευσης, πιστοποίησης όπως τα άλλα. Θα ήθελα την ε, προσέγγιση του θετικού καταλόγου, γιατί αυτό είναι καλύτερο για λόγους ρύθμισης, δηλαδή τι μπορεί να απελευθερωθεί και τι όχι, φαίνεται καλύτερα έτσι, με δυνατότητα μεγαλύτερης ασφάλειας και επίση ε, οι επιδοτήσεις για τον πολιτισμό, για τα μέσα, για εκπαιδευτικά ιδρύματα δεν θα ε, επηρεάζονται από αυτή τη συμφωνία και θα υπάρχει σαφής δυνατότητα να διατηρήσουμε τις δυνατότητες που έχουμε. Αν ε, περάσουν αυτά θα μπορέσουμε να περάσουμε την έκθεση από την Επιτροπή και να πάμε και στην Ολομέλεια ώστε να προβάλλουμε την απόψή μας για τη συμφωνία TTIP. Σας ευχαριστώ για τη σημαντική σας ε, ε, σταθερότητα. Κρατήσατε μια σταθερή γραμμή που συμφωνήθηκε μεταξύ των συναδέλφων. Αρχίζουμε αμέσως με την έκθεση της τροπολογία 14 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Περνάμε στην τροπολογία 15. Α, όχι, συγγνώμη, έχει αποσυρθεί. 22. 21 μάλλον. Γιατί 22 ήταν ταυτόσιμη. Α, 21 και 22 είναι ταυτόσιμες, υπέρ κατά αποχές έλεγχος. No, allora ho visto male, era, è scontrolliamo. Εγκρίνεται. Είδα λάθος. Πάντω δεν σηκώνετε τα χέρια σα και δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Σα παρακαλώ, ε, σηκώνετε τα χέρια σα 16. Υπέρ. Κατά. απόχέ. Εγκρίνεται. 17. Υπέρ. Κατά. απόχέ. Εγκρίνεται. 19. Τροπολογία 19. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 20 έχει αποσυρθεί. Πάμε σε συνδυαστική 2. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 26 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 27 ε, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 28 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 29 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 32. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 33. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 34. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 35. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 36 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 38 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 40 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 41 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 42 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 43 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 45 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 46 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 47 υπέρ Κατά αποχές απορρίπτεται. 48 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 50 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 51 υπέρ. Κατά αποχές γκρίνεται. 49 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Υπέρ, 52 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 53, α, με συγχωρείτε, 54 υπέρ κατά αποχές έλεγχος. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 55 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 56 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι απορρίπτεται. 57 υπέρ κατά <coughs> αποχές έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος της ψηφοφορίας εγκρίνεται 70 ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές νομίζω πως απορρίπτεται 61 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 62 ε, που είναι ταυτόσιμο ε, με την 63 και με την 64 και την 65 ΠΕΡ ε, κατά αποχές εγκρίνεται Περνάμε στην, στην 72. Ε, Γκυγιόμ. 72 Γκυγιόμ. Υπέρ κατά αποχές. Έλεγχος. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 73. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 74. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 75 υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε 75 ελέγχουμε την ε, ψηφοφορία τέλος ψηφοφορίας Καλά έκανα και έλεγξα. Για μια ψήφο έγινε δεκτή. Εγκρίθηκε. Περνάμε στην 76. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 77. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 77. Α, με συγχωρείτε, η 1. Η 1. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 2. Ε, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 3. Υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 6 υπέρ κατά έλεγχος άρχεται η ψηφοφορία κλείνει η ψηφοφορία εγκρίνεται με μία ψήφο διαφορά. Τροπολογία 6. Δηλαδή 7. Υπέρ, κατά, αποχές. Νομίζω δεν απορρίπτεται. Τροπολογία 1. Πώς Όχι, 8 που τροποποιείται από την προφορική 1. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 1. Υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται η 11 υπέρ παρακαλώ σηκώστε τα χέρια σας υπέρ λοιπόν κατά αποχές ε, απορρίπτεται 12 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται 13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Και περνάμε στην τελεϊκή ψηφοφορία με ηλεκτρονική ψηφοφορία παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με 24 ψήφους. Συγχαρητήρια κυρία Τρόπολη για αυτή τη σημαντική σας έκθεση. Τελειώσαμε με τις ψηφοφορίες. Finito in tempo, <laughs> lo dico eh, Και Τώρα, πριν να συνεχίσω, θα ήθελα να καλωσορίσω και στέφαμε προς τη συνάδελφο Ζούλη Γουόρντ, να καλωσορίσω τους φιλοξενούμενους της ε, κυρίας Γουόρντ, ε, που έρχονται από το Newcastle. Είναι μια οργάνωση που θέλει να δώσει μια εκπαίδευση του τσίρκου για, την, για τους νέους. Τσίρκο. Πού που κάνουν τέτοιου είδους ε, εργασία. Μπράβο. Ε, Έλεν και Άννα Τόμσον. Θα σας δώσω και τη διεύθυνση ενός αντίστοιχου σχολείου που φτιάχτηκε στην πόλη μου και δεν ξέρω για σας, αλλά σε εμά είναι περισσότερο τα κορίτσια που γράφονται σε αυτό το είδους τα μαθήματα. Πρέπει να το καταλάβουμε και λίγο αυτή τη δυναμική. Έχουμε τώρα την ανταλλαγή απόψεων με την Ευρώπη των φεστιβάλ. Φεστιβάλ για την Ευρώπη. ΕΦΕ λέγεται. Τα αρχικά είναι ΕΦΕ αυτή η Ευρώπη των φεστιβάλ για να ασχοληθούμε με το πρόγραμμα πιλότου που στηρίχθηκε τότε την εποχή του από την Επιτροπή Πολιτισμού. Ξεκίνησε το 2014. Α, συγγνώμη, μήπως μπορείτε να κάνετε λιγότερο θόρυβο. Ησυχία παρακαλώ, γιατί δεν είναι πολύ ευγενικό να κάνουμε θόρυβο για τον καλεσμένο μας. Σαμπίνα. Συγγνώμη Σαμπίνα. Γεια σας. Ευχαριστώ. Είχαμε βάλει λοιπόν αυτό το πρόγραμμα για τα φεστιβάλ ε, στον προϋπολογισμό μας για το 2014. Στόχος μας είναι ε, να μπορέσουμε διαχρονικά να δημιουργήσουμε μια πλατφόρμα για τους επαγγελματίες και για τους πολίτες, ώστε όχι μόνο να δικτυωθούν και να προωθηθούν, αλλά και για να βελτιωθεί η ποιότητα των φεστιβάλ το τομέα του πολιτισμού για να μπορούμε να αυξήσουμε την πρόσβαση στα διάφορα φεστιβάλ της Ευρώπης για τους καλλιτέχνες, για τις νέες παραγωγές αλλά και να δώσουμε ε, πληροφορίες κλειδιά για το τι συμβαίνει. Ποια είναι τα πολιτιστικά φεστιβάλ στην Ευρώπη. Έχουν δημιουργήσει δε και ένα πόρταλ ε, πολύ ενδιαφέρον. Εμείς έχουμε πολύ υπερασπιστεί ε, την, ευρωπαϊκή, ε, ε, την ευρωπαϊκή δημιουργία, την ευρωπαϊκή δημιουργικότητα. Το πόρταλ θα, πρέπει να, γίνει, να γνωστοποιηθεί περισσότερο και να δούμε και με ποιο τρόπο κυκλοφορεί η τέχνη και ο πολιτισμός στην Ευρώπη. Θα σας δώσω το λόγο. Ξέρω ότι έχουμε δύο υπεύθυνους που είναι σήμερα παρόντες. Θα δώσω το λόγο στην Κατρίν Ντεβέντερ που είναι γενική, γενική γραμματέας του φεστιβάλ και είναι παρόν και ο Ούγκο που είναι γενικό συντονιστή. στο Βέλγιο αλλά και διεθνώς. Παρακαλώ. Δεν είμαι συνηθισμένη να παίρνω το λόγο σε τέτοιες επιτροπές. Καλημέρα, ε, μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρία Πρόεδρε, πάντα είναι μεγάλη χαρά ε, να έχω τη δυνατότητα να απευθύνω το λόγο στους εκπροσώπους πολιτών από όλη την Ευρώπη. Πάντοτε είμαι πολύ συγκινημένη σε τέτοιες ε, εκδηλώσεις. Είμαι συνδιευθύντρια σε αυτό το πρόγραμμα μαζί με τον Ούγκο Ντεγκρέφ ε, που συνδιευθύνει και εκείνος. Να σας ευχαριστήσω καταρχήν που μας δώσατε χρόνο για να παρουσιάσουμε το πιλωτικό πρόγραμμα ΕΦΕ το οποίο αναπτύξαμε και αρχίσαμε μαζί με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και θέλουμε να κάνουμε μια ανασκόπηση του προγράμματος και να πείσουμε όπως ελπίζουμε τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι αξίζουν περαιτέρω επενδύσεις εδώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε διανύμει και υλικό που ελπίζω ότι θα σας δώσει ακόμη περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα. Όπως είπε η Σίλβια Κώστα, η πρόεδρος της Επιτροπής, συμφωνούμε ότι η Ευρώπη είναι ήπειρος φεστιβάλ, ε, μεγάλα, μικρά, στο βορρά, στο νότο, ανατολή, δύση, σε μικρές πόλεις, μεγάλα φεστιβάλ. Φεστιβάλ υπάρχουν σε κάθε γωνιά της Ευρώπης. Τα φεστιβάλ ε, γίνονται εδώ και αιώνες ολόκληρη την Ευρώπη και στις πόλεις και στην Ήπεθρο συνενώνουν σε μια εορταστική ατμόσφαιρα τους ανθρώπους. Εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση Φεστιβάλ πάνω από ε, έξι χρόνια έχουμε εμπειρία και ξέρουμε ότι τα φεστιβάλ ε, εμπλουτίζουν τα πολιτιστικά δρόμενα. Ε, είναι σημαντικό να ξέρει κανείς ποια φεστιβάλ κάνουν την πιο καινοτόμο και ενδιαφέρουσα δουλειά. Επίσης είδαμε ότι υπάρχει ανάγκη μιας συμμαχίας ε, ε, των φεστιβάλ που έχουν παρόμοιους ε, στόχους. Έχουμε ένα ε, πολιτιστικό χώρο που θέλουμε να είναι γνωστός. Τα φεστιβάλ είναι σημαντικές στιγμές πολιτιστικές, καλλιτεχνικές που συνενώνουν τους πολίτες επί ευρωπαϊκών αξιών θέλω με τα φεστιβάλ, ε, εταίροι να αναπτύξουν τις δραστηριότητες αυτές περισσότερο. Τι έχουμε επιτύχει μέχρι τώρα. Είναι σημαντικό να ξέρετε ποια βήματα ε, κάναμε μαζί για την πλατφόρμα, ε, για τα ευρωπαϊκά φεστιβάλ, τη, ε, μαζί με, με τα θεσμικά όργανα. Το 2010 το πολιτιστικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής άρχισε να έχει και ένα τμήμα για φεστιβάλ. Ήταν πολύ φιλόδοξο και βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Είχε όμως περιορισμένες δυνατότητες γιατί οι δικαιούχοι που επελέγησαν ήταν πολύ λίγοι. Στο πρόγραμμα είχε δοθεί μια επιδότηση περιορισμένη σε μικρό αριθμό φεστιβάλ. Για παράδειγμα, 674 ε, ε, φεστιβάλ ζήτησαν επιδότηση και μόνο 18 επελέγησαν το 2010. Το 12, 235 φεστιβάλ έκαναν αίτηση. Αυτό δείχνει μειούμενο ενδιαφέρον από την πλευρά των φεστιβάλ επειδή το ποσοστό επιτυχίας ήταν πολύ μικρό. Και μπορούμε να συμπεράνουμε επίσης ε, ότι έτσι ήταν λίγο, ε, ε, ε, περιορίστηκε το ευρωπαϊκό αυτό πρόγραμμα. Ενώ αν ήταν αλλιώ τα πράγματα, πολλοί θα ήθελαν να το προωθήσουν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αντέδρασαν σε αυτή τη μείωση του ενδιαφέροντο και άρχισαν ένα πιλωτικό πρόγραμμα για την πλατφόρμα και φεστιβάλ καλλιτεχνικά. Αφού αναπτύχθηκε αυτή η ιδέα μαζί με την ΕΦΑ, την Ένωση ε, και στη συνεργασία με τον πρόεδρο Ντάρκο Μπούλε και με τον Νου Βεντεγκρέφ και βέβαια είχα και εγώ το προνόμιο να παρουσιάσω αυτή την ιδέα το 2011 στην Ευρωπαϊκή ε, ε, Επιτροπή, Πολιτισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, μετά ανατέθηκε στην ΕΦΑ να εφαρμόσει το πιλωτικό πρόγραμμα. Η ΕΦΑ επελέγει από, ανάμεσα από πολλούς ετούντες. Ε, μαζί με, το πρόγραμμα, την ε, ε, μονάδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το πολιτι... υπεύθυνη για το πολιτιστικό πρόγραμμα ε, αναπτύσσουμε τώρα το ΕΦΕ ε, μέσα από συνεχιζόμενη συνεργασία. Το πιλωτικό πρόγραμμα παρουσιάστηκε και συζητήθηκε και με τον ε, Πίτροπο Ποτιμπορνάβροτσης και έγινε δεκτό. Ε, η κυρία Κώστα, η πρόεδρος, επίσης υποστήριξε το πρόγραμμα ΕΦΕ που είπατε ήδη ότι καταδεικνύει την, ε, το δυναμικό των τεχνών και του πολιτισμού. Ε, έτσι προωθούνται φεστιβάλ που εμπλουτίζουν όχι μόνο τα ίδια τα φεστιβάλ αλλά τους καλλιτέχνες και τους πολίτες διότι Έχουμε ε, και πλατφόρμα online, ένα ε, σήμα και έτσι μπόρεσαν ε, μέσα από ένα πρόγραμμα labeling να εγκριθούν πολλά φεστιβάλ. Τώρα θέλουμε να φτάσουμε σε ακόμα μεγαλύτερο αριθμό φεστιβάλ. Ήδη 600 παραλήπτες του σήματος υπάρχουν και επηρεάστηκαν ε, αν και ήταν ε, μικρό ε, το ποσό που έλαβαν, ο αριθμός των φεστιβάλ που οργανώθηκαν και υπέβαλαν αίτηση έφτασε στον αριθμό των 1666, που είναι σημαντικό. βλέπουμε λοιπόν ανάπτυξη, αύξηση του ενδιαφέροντος και πολλά φεστιβάλ αφιέρωσαν χρόνο για να ζητήσουν υποστήριξη οικονομική από την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ε, ήταν και μικρή. Τι πετύχαμε λοιπόν στο πρώτο δωδεκάμινο λειτουργίας αυτού του πιλωτικού προγράμματος. Μπορούμε να σας πούμε ότι 897 ε, φεστιβάλ έκαναν αίτηση, 31 χώρες συμμετέχουν στην πλατφόρμα, όλα τα 28 κράτη-μέλη, συν 3 μη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, πολλά φεστιβάλ ετούντα θα καταλήξουν σε ποιοτικό σήμα, περίπου 10 θα ε, βραβευθούν ε, Οχτώ προσωπικότητες σε υψηλού κύρους συμμετέχουν στην Κριτική Επιτροπή των Φεστιβάλ. 24 κέντρα φεστιβάλ ε, ε, δημιουργήθηκαν με εθνικούς αντιπροσώπους που εργάστηκαν για να προωθηθούν τα φεστιβάλ σε εθνικό επίπεδο. Σε κάθε νέα χώρα δημιουργείται ένα κέντρο φεστιβάλ που είναι το τοπικό σημείο επαφής, σύνδεσμος δηλαδή έγιναν αξιολογήσεις σε εθνικό επίπεδο των αιτήσεων ήδη από τα κέντρα. Ε, τώρα θα δημοσιευθεί και ένα βιβλίο εμπνεύσεων το οποίο θα εμβαθύνει στο τομέα των φεστιβάλ και θα παρουσιάσει τα φεστιβάλ που έχουν το σήμα και το, πήραν και το βραβείο ΕΦΕ. Ε, όλα αυτά θα παρουσιάζονται και σε πλατφόρμα online και έτσι θα έχουν μεγαλύτερη πρόσβαση στην πολιτιστική ε, πολυμορφία οι πολίτες. Επίσης ε, θα γίνει εορτασμός ε, για να, με τη συμμετοχή των βαρδευθέντων. Το 2015 το πρόγραμμα θα προωθηθεί διεθνώς προβάλλοντας την Ευρώπη ως πολιτιστική προ... ήπειρο σε όλο τον κόσμο. Όλα αυτά θα γίνουν από τον Ιούνιο μέχρι το τέλος του χρόνου. Ε, μαζί μπορούμε να φροντίσουμε οι δραστηριότητες αυτές να συνεχιστούν ε, ικανοποιητικά και στο μέλλον. Ε, ο αριθμός των φεστιβάλ είναι απεριόριστος ε, και μπορεί να προωθηθούν πολλά από αυτά μέσω χάρη στη συνεχιζόμενη συνεργασία μας πώς θα προχωρήσουμε στο μέλλον. Νομίζω ότι από κοινού πρέπει να δούμε πώς το project θα συνεχιστεί στα πλαίσια των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Γι' αυτό το λόγο ε, έχω την ευκαιρία και το προνόμιο να σας απευθύνω το λόγο σήμερα, να εντάξω το θέμα στο χρονοδιάγραμμά σας και να συζητήσουμε τη φάση 2 μια επόμενη διετία του προγράμματος ώστε να αναπτύξει το πλήρες δυναμικό του. Περισσότερες λεπτομέρειες. Η πλατφόρμα όπως είπα καλύπτει όλη την Ευρώπη και ε, έχει πάρα πολλά σημαντικά θέματα. Ε, είναι απλή η δομή του. Ε, στη δημιουργική Ευρώπη η ΕΦΑ αποτελεί μια πλατφόρμα. Στα μάτια τα δικά μας αυτό σημαίνει ότι η ΕΦΑ είναι μια κοινότητα είναι η νέα κοινότητα των φεστιβάλ που συγκεντρώνει φεστιβάλ από όλα τα είδη, από όλα τις τέχνες και τις ε, πολιτιστικές δραστηριότητες με ρίζες στην τοπική κοινότητα ε, και με ε, δρόντες ευρωπαϊκούς και παγκόσμιους. Αυτά είναι τα τρία κριτήρια που προωθήσαμε στο, στην πρώτη φάση. Η αποστολή μας μπορεί να περιγραφεί ε, με τις λέξεις γιορτάζουμε και εμπλουτίζουμε. Ε, τιμούμε τα πιο σημαντικά φεστιβάλ τεχνών και πολιτισμού. Η πλατφόρμα διασφαλίζει ένα σχήμα ποιότητας για τα ευρωπαϊκά φεστιβάλ και επίσης και ένα βραβείο για το... Όλα τα φεστιβάλ εορτάζονται σε έναν οδηγό φεστιβάλ online. Θα είναι ελεύθερης πρόσβασης για τους πολίτες όλης της Ευρώπης και όλου του κόσμου επίσης. Έτσι μπορούν να ανακαλύπτουν οι ε, πολίτες ε, τα πιο ενδιαφέροντα φεστιβάλ. Η πρόσβαση δεν έχει εξασφαλιστεί ακόμα, αν και ξέρουμε ότι η Ευρώπη είναι ήπειρος των φεστιβάλ. Ε, δεν υπάρχει κεντρική τοποθεσία, ε, κεντρικός τόπος. Τώρα με τον οδηγό θα μπορούμε να έχουμε αυτή τη δυνατότητα για να προβάλλονται στους Ευρωπαίους και σε όλο τον κόσμο οι αξίες που υιοθετεί και προβάλλει η Ευρώπη. Η ΕΦΑ επίσης εμπλουτίζει, εμπλουτίζει το τοπίο των φεστιβάλ διότι προωθεί τάση στην καλλιτεχνική αριστεία και την καινοτομία στα φεστιβάλ. Η πλατφόρμα θέλει να διευρύνει την ε, γνώση του τι συμβαίνει, ε, να προωθήσει την καινοτομία και την αριστεία. Εμείς έχουμε και μια ψηφιακή πύλη, ε, μπορεί έτσι να υπάρξει ανταλλαγή ψηφιακά γνώσεων, πληροφοριών, προβάλλοντας το τοπίο των φεστιβάλ. θα, τα φεστιβάλ βεβαίως φέρνουν κοντά όλους όσους εργάζονται ή ενδιαφέρονται για τα φεστιβάλ. Ε, τους διευθυντές, ε, τους ε, δρόντες, παράγοντες κλπ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εγγυάται την εξαιρετική ποιότητα. Όλοι θα ωφεληθούν από μια αυξημένη ορατότητα, συμμετοχή των φεστιβάλ στην καλλιτεχνική κοινότητα και την αναγνώριση των καλλιτεχνικών εξαιρετικών αξιών το επόμενο βήμα θα είναι η εξέλιξη του τοπίου για τα καλλιτεχνικά και πολιτιστικά φεστιβάλ. Για να επιτύχουμε την αποστολή μας προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε ισχυρή συμμαχία εταίρων σε όλη την Ευρώπη. Η ιδέα του ΕΦΕ δεν είναι από πάνω προς τα κάτω αλλά από κάτω προς τα πάνω. Η ΕΦΕ λειτουργήσε σε συνεργασία όπως είπα με κέντρα φεστιβάλ, οι εθνικοί εκπρόσωποι, ε, τους εθνικούς εκπροσώπους δηλαδή σε 24 χώρες. Αυτά τα κέντρα είναι ένα ε, στοιχείο ε, σημαντικό, αποκεντρωτικό. Ε, υπάρχουν ε, νέοι που γνωρίζουν το τοπίο επιτόπου που συνδυάζουν τις προσπάθειες όλων των ενδιαφερομένων και στη χώρα τους και σε όλη την Ευρώπη ε, για να προωθηθεί το καινοτόμο αυτό πρόγραμμα. Στο μέλλον ελπίζουμε όλα τα κράτη-μέλη να εκπροσωπούνται με κέντρα όπως και άλλες γειτονικές χώρες που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη και να συμμετέχουν και σε αυτά την πλατφόρμα των Φεστιβάλ ΕΦΕ με αυτή την πανευρωπαϊκή διαδικασία τα, τα καλύτερα φεστιβάλ ε, θα βραβευτούν και θα πάρουν το σήμα. Οι αιτήσει άρχισαν το καλοκαίρι του 2014, έκλεισα το Δεκέμβριο και οι εμπειρογνώμονες ε, που επελέγησαν από τα κέντρα εξέτασαν τις αιτήσει. Ε, υπάρχουν τώρα 100 προσωπικότητες, κριτικοί, δημοσιογράφοι, οργάνωτες, φεστιβάλ, καλλιτέχνες κλπ. που συμμετέχουν στην Κριτική Επιτροπή και εργάστηκαν στα πλαίσια αυτής της πλατφόρμας. Και αυτό ήταν πολύ επιτυχές. Εκτός από τα κέντρα και τους ειδικού και εμπειρογνώμονες, ε, δημιουργήθηκε και μια επιτροπή του φεστιβάλ, ομάδα δηλαδή ε, ατόμων από όλη την Ευρώπη που θα λάβουν την τελική απόφαση για τα φεστιβάλ που θα πάρουν το σήμα και τα φεστιβάλ που θα ε, είναι υποψήφια για βράβευση. Έχουμε τον διευθυντή που εδρεύει στη Λοζάνη τώρα και ήταν ο πρώην διευθυντής του Φεστιβάλ της Αβινιών. Ε, υπάρχουν διευθυντές φεστιβάλ που συμμετέχουν, ε, η Ορτάντσα ε, Σνεβούρ, στην Διευθύντρια, ο Τόμ Κρίτ, Διευθυντής Όπερας, ο Πιέτρου Κοζίνσκι, δραματουργός από την Πολωνία, Ούλρικε Γιώζεψον, καλλιτεχνικός διευθυντής στο Γκέθεμπορκ Νίνα Πέτς, διευθύντρια του Κινηματογραφικού Φεστιβάλ, ε, και πολλοί άλλοι από τη Νέα Υόρκη, ο Γιώργη Σάμπο, ε, διευθυντής του House of Contemporary Art ε, στη Βουδαπέστη. Η ΕΦΑ λοιπόν, η ΕΦΕ θέλει ισχυρού εταίρου για να έχουμε καλά αποτελέσματα σε πολλά επίπεδα. Οικοδόμησε πάνω στο υπάρχον δίκτυο της, του συνδέσμου ή της Ένωσης των Φεστιβάλ των, της Ευρώπης, θέλω να αναφέρω κάτι ακόμα. Υπάρχει ένας εκδοτικός οίκος με τεράστια πείρα στον καλλιτεχνικό τομέα και ανέλαβε να δημιουργήσει τον καλλιτεχνικό οδηγό και τον οδηγό των φεστιβάλ. Υπάρχουν πολλές συνεργασίες στον ψηφιακό κόσμο που θα ακολουθήσουν στο μέλλον. Αυτή τη στιγμή είμαστε στα μέσα της διαδικασίας του προγράμματος, οπότε μόνο τα ε, επιτεύγματα μέχρι τώρα μπορώ να παρουσιάσω. Βλέπετε, ελπίζω, ότι υπάρχουν ε, πολλά ωφέλη από το πρόγραμμα αυτό. Τώρα υπάρχουν ορισμένα στοιχεία ε, όπως ε, η Διεθνής Επιτροπή που, των φεστιβάλ που θα λάβει τελική απόφαση για το σήμα και την, ε, τα βραβεία, τα φεστιβάλ που θα προωθηθούν αφού θα πάρουν το σήμα, θα γίνει επίσης η έκδοση του οδηγού, η δημοσίευση του έκδοση του βιβλίου και η ορταστική εκδήλωση ε, το Σεπτέμβριο φέτος το 2016. Ελπίζω ότι θα αρχίσω με την ετήσια διαδικασία αυτή πάλι από την αρχή, αλλά γι' αυτό όπως είπα και πριν χρειαζόμαστε τη συνεχιζόμενη υποστήριξή σας για να χτίσουμε πάνω στην επιτυχία που είχαμε μέχρι τώρα. Καθώς μεγαλώνει το πρόγραμμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση των Φεστιβάλ ως οργάνωση και ως δίκτυο των φεστιβάλ θα συνεχίσει να στηρίζει το project με τα μεγάλα δίκτυα και σημαντικούς εταίρους της θα, εμείς θα δράσουμε ως πυρήνας ενεργός ε, που θα έχει συγκεντρώσει γνώση για τα φεστιβάλ ε, και έτσι θα επεκτείνουμε την πλατφόρμα των φεστιβάλ. Η ΕΦΑ προσφέρει το δίκτυό της ε, ούτω ώστε να αντλήσουμε περισσότερη δημιουργικότητα από τα φεστιβάλ. Η ΕΦΗ είναι το αποτέλεσμα πολυετού συνεργασίας μεταξύ Κομισιών και Κοινοβουλίου εδώ στις Βρυξέλλες χάρη στο ε, στην παρελθούσα και τωρινή εργασία της ΕΦΑ νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2013 ε, δικαίως ανέθεσε στην ΕΦΕ να δημιουργήσει την πλατφόρμα αυτή που θα κάλυψε ένα διάστημα διετές. Η ΕΦΑ είναι έτοιμη να συνεργαστεί σε στενή συνεργασία όπως και στο παρελθόν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να συζητήσει πώς το πιλωτικό πρόγραμμα θα συνεχίσει για να βελτιώνει την οργανωτική του δομή και να αυξάνει τον αντίκτυπο που θα έχει μακροπρόθεσμα. Οι προσπάθειες και τα αποτελέσματα μέχρι τώρα από την πρώτη φάση πρέπει να συνεχιστούν με τη δομή που δημιουργήσαμε. Για να είμαστε βιώσιμοι, πιστεύουμε το πρόγραμμα αυτό έχει μακροπρόθεσμα δυναμικό να είναι το κέντρο της ζωής των φεστιβάλ στην Ευρώπη. Τα φεστιβάλ ε, συμπεριλαμβάνουν πολλούς ανθρώπους, καλλιτέχνες, διευθυντές ε, κλπ. Είναι λοιπόν ε, ένας κλάδος σημαντικός και οι επενδύσεις εκεί θα έχουν απόδοση διότι όλοι αυτοί οι δρόντες θα μπορούν να βελτιώσουν το ευρωπαϊκό project και τις αξίες που προβάλλει. Ε, όλα αυτά τα χρόνια οι επιτυχίες ήταν πολλές. Όλοι οι εμπλεκόμενοι που προανέφερα αποτελούν τώρα μέρος αυτής της πλατφόρμας. Ε, θέλουν και ελπίζουν ότι θα δοθεί συνέχεια για να συνεργαστούμε όλοι μαζί για να εμπλουτίσουμε και να ερωτάσουμε τον τομέα των φεστιβάλ. Ε, τελειώνω λέγοντας ε, ότι είμαστε βέβαιοι ότι βλέπετε τις αξίες ε, που ενέχονται εδώ και τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ελπίζω ότι θα, μπορέσουμε, θα μπορέσουν να εγκρίνουν τον συντονισμό του πιλωτικού προγράμματος όταν περάσουμε στις επόμενες φάσεις συνέχισης του. Ε, και από τον επόμενο προϋπολογισμό. Τα μέλη της Επιτροπής Πολιτισμού και πρόεδρος, ε, ε, μέλη της Επιτροπής Πολιτισμού, πρόεδρε κυρία Σίλβια Κώστα, ευχαριστούμε για την πρόσκληση και είμαστε στη διάθεσή σας για να απαντήσουμε σε τυχόν ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή σας την εισήγηση και επειδή αφηνήσατε, την έννοια και την προοπτική αυτής της πλατφόρμας που στόχο έχει να στηρίξει και να, την κυκλοφορία των καλλιτεχνών σε ολόκληρη την Ευρώπη, αλλά και να προωθήσει ένα είδος <clears throat> σήματος ποιότητας για τα φεστιβάλ αυτά που έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Πιστεύω ότι αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα απέδειξε ότι είναι πολύ, ε, ότι εκτιμάται ιδιαίτερα όταν ε, βλέπουμε πόσοι ε, ε, ζητούν πληροφορίες. Ε, τα, αυτοί οι κόμβοι θα έπρεπε να ενισχύσουν και ίσως να μας δώσετε πληροφορίες και εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το πώς λειτουργούν. Γι' αυτό θεωρούσα, θεώρησα ε, χρήσιμη αυτή την ανταλλαγή απόψεων Λοιπόν, Τρούπελ, Βόρντ και Σετροϊβά έχουν ζητήσει το λόγο. Αν υπάρχουν και άλλα, μου το πείτε. Ευχαριστώ πολύ για την ενδιαφέρουσα παρουσία σας. Θα ήθελα να μου πείτε εάν είχατε προβλήματα με, για την δημιουργία αυτής της πλατφόρμας. Εάν υπάρχουν προτάσεις για βελτίωση και αν ναι, ποιες είναι προτάσεις. Η ευχαριστώ πολύ για την παρουσίασή σας. Εγώ είμαι υπέρμαχος τέτοιου είδους ε, φεστιβάλ, διότι πρόκειται για ένα τρομερό ε, εορτασμό του κουλτούρας του καθενός και μεγάλη ευκαιρία. Θα ήθελα όμως να κάνω μία ε, προειδοποίηση. Δεν θα πρέπει να γίνεται κάτι σε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο ώστε να αποκλείονται κάποιοι οι οποίοι είναι πάρα πολύ καλοί σε τοπικό επίπεδο. Θα πρέπει λοιπόν να είστε αντικειμενικοί σε όλα. Θα ήθελα να μου πείτε πώς μετράτε την ποιότητα ε, και το ακροατήριο μπορεί να εκφράσει επί αυτού του θέματος νόμι. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει όντως να προωθήσουμε ό,τι είναι τοπικό και να είμαστε συγκεντρωτικοί και να συμπεριλαμβάνουμε τους πάντες αντί να αποκλείουμε τον οποιοδήποτε. Ευχαριστώ. Κυρία ευχαριστώ πολύ. Πάντα καλό είναι να βλέπει κανείς ένα πιλωτικό πρόγραμμα και χαίρομαι που έχουμε μία πλατφόρμα που μπορεί να προωθήσει τα φεστιβάλ. Θα πρέπει όμως να ξέρουμε ότι ένα πιλωτικό πρόγραμμα είναι ένα πιλωτικό πρόγραμμα το οποίο έχει την, ε, το χρόνο ζωής του, την αρχή του και το, και το τέλος του. Εάν πρέπει να έχουμε ένα κονδύλι για να χρηματοδοτούνται τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Μπορείτε να μας πείτε γιατί κονδύλι θα πρέπει να μιλάμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για αυτή την πρωτοβουλία, η οποία κατά την άποψή μου είναι εξαιρετικά σημαντική, διότι επιτρέπει να έχουμε και ποιοτικέ πληροφορίες για τα διάφορα φεστιβάλ που οργανώνονται στην Ευρώπη. Αν δεν με πατάει η μνήμη μου, πάρα πολλά φεστιβάλ οργανώνονται στην Ευρώπη. 7 με 10.000 αν δεν κάνω λάθος. Βεβαίως υπάρχουν πάρα πολλοί γνωστά φεστιβάλ όπως το φεστιβάλ Mozart στο Salzburg, φεστιβάλ θεάτρου όπως τη Σαββινιό ή του Εδιμβούργου. Έχουμε λοιπόν πολλές πληροφορίες για αυτά τα παραδοσιακά και πολύ γνωστά φεστιβάλ. Επίσης, υπάρχουν φεστιβάλ τα οποία είναι πάρα πολύ δαπανηρά. Για τα οποία ζητείτε σημαντική χρηματοδότηση χωρίς να έχουν ε, ποιότητα τελικά. Είναι σημαντικό λοιπόν να έχουμε την κατάλληλη ενημέρωση για τα διάφορα φεστιβάλ και την ποιότητά τους. Εγώ ίδιος πρέπει να πω ότι έχω επισκεφθεί περισσότερα από 500 φεστιβάλ στην Ευρώπη. Βλέπω πώς εξελίσσονται και μπορώ να πω ότι ακόμη και αν ένα φεστιβάλ είναι ποιοτικό δεν σημαίνει ότι θα παραμείνει για πάντα ποιοτικό. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Αυτό είναι ένα από τα προβλήματα που πρέπει να εξετάσουμε στην Ευρώπη. Επίσης, πρέπει να πω ότι γίνονται διάφοροι επαιτειακοί εορτασμοί στην Ευρώπη, αλλά τα φεστιβάλ διεξάγονται κάθε χρόνο σχεδόν και μια εξαιρετική ευκαιρία για να προωθήσουμε τις ευρωπαϊκές αξίες. Ευχαριστώ. δεν υπάρχουν άλλοι συνάδελφοι που ζητούν το λόγο, θα ήθελα δώσω τον Καρέλ Μπαρτάκ, εκπρόσωπο της Επιτροπής των Ευχαριστώ που εδώ. Ευχαριστώ σας, ευχαριστώ Πρόεδρε. Εδώ αναφέρθηκε η σπουδαιότητα αυτών των φεστιβάλ για την κουλτούρα της Ευρώπης, που όλο και περισσότερο μεγαλώνει. Και Βλέπουμε έτσι τι σημαίνει κουλτούρα και πολιτισμός για τις ε, διαφορετικές χώρες της Ευρώπης. Τα φεστιβάλ λοιπόν αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά για την ε, κουλτούρα και της Ευρώπης και την πρόθεση της. Είναι σημαντικά τέτοιου είδους ε, φεστιβάλ, η πλατφόρμα αυτή είναι σημαντική διότι έτσι μπορούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο να κατανοημίσουμε καλύτερα περί τίνος πρόκειται και να μπορέσουμε στους πολίτες των διαφορετικών χωρών της Ευρώπης να παρέχουμε την κατάλληλη πληροφόρηση για το τι γίνεται και εκτός των συνόρων της ε, κάθε χώρας του καθενός και ποιες είναι οι δυνατότητες παρακολούθησης. Παρακολουθούμε τους είναι σε αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα από την αρχή της δημιουργίας και μπορώ να πω μετά από ένα χρόνο ύπαρξη αυτού του πολιτικού, του πιλωτικού προγράμματος ότι μετά από κάποιους ενδιασμούς βλέπουμε ότι πραγματικά διαφοροποιείται τώρα σε, στην Ευρώπη σε σχέση με ό,τι άλλο υπάρχει σε επίπεδο φεστιβάλ. Ακούσατε τους αριθμούς, είδατε ότι υπάρχουν περίπου 9.000 φεστιβάλ τα οποία συμμετέχουν, έχουμε τα hubs αυτά, τους, τα κομβικά κέντρα και τα αποτελέσματα του πρώτου ετούς ανταποκρίνονται στις προσδοκίες του πιλατικού ε, σχεδίου αυτού. Τώρα, θα έχουμε την ε, δεύτερη χρονιά του πιλωτικού αυτού σχεδίου και αναμένουμε <laughs> ότι θα επεκταθεί και θα, γίνουν, θα παγιωθούν ακόμη περισσότερο σε ευρωπαϊκό επίπεδο και θα πρέπει με την ε, ένωση των ευρωπαϊκών φεστιβάλ να δούμε πώς θα εξελιχθούν, πώς θα αναπτυχθούν περαιτέρω. Όπως ελέγχθη, κάτι πιλωτικό είναι πιλωτικό, έχει αρχή και τέλος. Και θα πρέπει να δούμε πώς θα συνεχίσουμε, αν θα συνεχίσουμε με αυτό τον τρόπο, αν θα επεκταθεί αυτή η δράση, ούτως ή άλλως η Ένωση των Φεστιβάλ της Ευρώπης προσπαθεί να μελετήσει το πώς θα εξελιχθεί το πρόγραμμα αυτό, το project αυτό, ώστε να ε, μπορέσει να ανταποκριθεί στις ε, πολιτιστικές προτεραιότητες που υπάρχουν, αν θα έχει ναι, καινοτόμο, αν θα μπορέσει συμπεριλάβει ε, μικρά πολιτιστικά σχέδια, αν θα μπορέσει να επωφεληθεί από τι εξελίξει τη ψηφιακή τεχνολογία. Όλα αυτά είναι σημαντικά ώστε να μπορέσει να γίνει βιώσιμο το όλο σχέδιο και σε μερικά χρόνια θα πρέπει να δούμε πώς έχει εξελιχθεί και εάν θα αποτελέσει αναπόσπαστο μέλος της ε, προσπάθειας των πολιτιστικής που γίνεται σε όλη την Ευρώπη. Ούτως ή άλλως πρέπει να πω ότι για μας υπάρχει η δυνατότητα, ανήθευση στις δυνατότητες, πώς μπορούμε να προωθήσουμε την κινητικότητα των καλλιτεχνών, των νέων, που θα μπορούν ενδεχομένω να μετακινούνται από το ένα φεστιβάλ στο άλλο. Αυτό είναι μέρος του άλλου σχεδίου. Επίσης, εξετάζουμε τις δυνατότητες πρόθεσης και ανάπτυξης του καλλιτεχνικού τουρισμού. Διότι πρόκειται για κάτι το πολύ σημαντικό. Πρέπει να ξέρουν οι πολίτες τι γίνεται στην Ευρώπη και να μπορούν να μετακινούνται αναλόγως για να παρακολουθούν τέτοιου είδους φεστιβάλ. Γιατί υπάρχει ζήτηση. Πιστεύουμε ότι αξίζει να συνεχιστεί η προσπάθεια αυτή. Θα εργαστούμε περαιτέρω με το σχέδιο αυτό και θα δούμε επίσης όταν τελειώσει η πιλωτική φάση αυτή πώς μπορούμε να προσαρμόσουμε το σχέδιο αυτό σε συνθήκες οι οποίες θα άπτονται των ε, δημιουργικών πολιτιστικών δυνατοτήτων που έχουμε στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την Επιτροπή. Θα ήταν ενδιαφέρον να ακούσουμε τις απαντήσεις σας στις ερωτήσεις των συναδέλφων, ιδιαίτερα ε, τα κριτήρια ποιότητας και φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν διάφοροι προβληματισμοί, τα υποτιθέμενα σήματα όπως αποκαλούνται για όσους έχουν διεθνεί ε, βλέψεις, αλλά μην ξεχνάμε και τα πολιτιστικά, τα μικρά φεστιβάλ που ίσως να μην είναι διεθνού συμβελνικούς αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ποιοτικά. Έπειτα έχουμε ε, φεστιβάλ ε, βιβλίων, φεστιβάλ σινεμά, ε, τα ελαμβάνετε όλα υπόψη. Υπάρχουν πλευρές που σας απασχολούν περισσότερο, ή που περισσότερο άλλα, άλλες πτυχές. Ε. Έπειτα, στη χώρα μου υπάρχει κάτι, ένας άλλος προβληματισμός που είναι ενδιαφέροντας ε, και ή συγκεντρώνονται, μάλλον ε, φεστιβάλ ε, του πνεύματος, της φιλοσοφίας, της οικονομίας ανάλογα με την πόλη και είναι ε, πόλεις οι οποίες έχουν υιοθετήσει το θέμα αυτό για κάθε χρόνο και κάθε χρόνο δίνουν μια διεθνή διάσταση προβληματισμού σε αυτά τα θέματα χρησιμοποιώντας και πολιτιστικό και καλλιτεχνικό περιεχόμενο αλλά φαντάζομαι πως τοποθετούνται μέσα σε μια διάσταση πολιτιστική περισσότερο. Θα ήθελα να γνωρίζω λοιπόν αν έχετε υπόψη και αυτές τις περιπτώσεις. Ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις σας. Θα προσπαθήσω να απαντήσω μία προς μία, όχι, όχι με τη σειρά, αλλά με βάση τη σπουδαιότητα για το φεστιβάλ και το τι είναι ποιότητα και ποια είναι και τα κριτήρια της πλατφόρμας όχι μόνο της πλατφόρμας μάλιστα, αλλά και άλλα κριτήρια αξιολόγησης και αξιοποίησης των φεστιβάλ, καλλιτεχνικών φεστιβάλ. Κάνατε μια ερώτηση για την ποιότητα και μια ερώτηση για τον ορισμό, που άπτεται και τις ερωτήσεις σχετικά με τα προβλήματα και τις βελτιώσεις. Γιατί η πρώτη πρόκληση είναι να δώσουμε ένα ορισμό στο φεστιβάλ. Υπάρχουν πολλοί ορισμοί που έχουν σχέση με το ιστορικό υπόβαθρο ή το πολιτιστικό υπόβαθρο ε, ή το περιεχόμενο. Ε, ο δικός μας ορισμός είναι ότι το φεστιβάλ περιορίζεται σε χρόνο και χώρο συγκεκριμένο ότι ε, είναι μια γιορτή η οποία εξυπηρετεί την ε, πολιτιστική και καλλιτεχνική ανάπτυξη μιας κοινότητας, δηλαδή η, η, η καλλιτεχνική και πολιτιστική διάσταση είναι σημαντική σε ένα συγκεκριμένο χώρο και χρόνο. Ε, μια άλλη βάση μας είναι η συμμετοχή των, ε, των κοινοτήτων, ε, προβολή δηλαδή τους πολίτες σε ένα συγκεκριμένο χώρο, η οποία γίνεται πάνω στη βάση μια, ενός οράματος ε, καλλιτεχνικού ε, με δυνατότητα όμως προβολής και σε ευρύτερου χώρους. Δηλαδή μπορεί να είναι σε μια μικρή πόλη της ε, Φιλανδίας και να έχει προβολή ε, και βεβαίως από την άλλη έχουμε και μεγάλα καλλιτεχνικά του Εδιμβούργου που και αυτά πρέπει να προβάλλονται. Ή μεγάλα φεστιβάλ όπως τα Berliner Festspiele κλπ. Ε, οι κλίμακες δηλαδή μπορεί να είναι διαφορετικές, αλλά η πρόθεση θα πρέπει να γίνεται και τρίτον θα πρέπει το φεστιβάλ να ανταποκρίνεται σε μια να, να λειτουργήσει ευρωπαϊκή αλλά και παγκόσμια διάσταση. Αυτό μπορεί να εκφράζεται με διαφορετικούς τρόπους. Δεν είναι μόνο το ποσοτικό στοιχείο, όπως ας πούμε ο αριθμός των συμπαραγωγών μεταξύ διαφόρων χωρών, αλλά και τα θέματα είναι σημαντικά, αυτά που απασχολούν τα φεστιβάλ. Μπορεί να είναι πολύ τοπικά, περιορισμένα στο θεματολόγιο, που αφορούν περιβαλλοντικά θέματα, ε, για παράδειγμα, ε, ή άλλα θέματα πιο ε, ευραία. Υπάρχουν πολλές συνιστώσεις που πιστεύουμε ότι θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται σε κάθε φεστιβάλ, με διαφορετικό τρόπο όμως μπορούν να αντιμετωπίζονται και να προβάλλονται. Έτσι η ευρωπαϊκή διάσταση ε, μπορεί να ενταχθεί στα φεστιβάλ. Και αυτό είναι δύσκολο γιατί τα φεστιβάλ δεν είναι μόνο καλλιτεχνικά, δεν αφορούν μόνο χορό, θέατρο, ε, κινηματογράφα, δηλαδή υπάρχουν και φεστιβάλ που αφορούν φιλοσοφία, φιλοσοφικές συζητήσεις για το σημερινό κόσμο, αφορούν την ποίηση, τη λογοτεχνία. Ε, δεν υπάρχει αποκλεισμό κάποιων φεστιβάλ που λειτουργούν σε πιο εμπορική βάση. Ε, δεν αποκλείομαι δηλαδή τα φεστιβάλ rock, pop, κινηματογράφου, γιατί πιστεύουμε ότι η γνώση, ε, οι γνώσεις που αποκτούνται από τον έναν ε, προς τον άλλον ε, είναι πολύ σημαντική και σε αυτού του είδους τα φεστιβάλ. Πάνω απ' όλα μας ενδιαφέρει να δημιουργήσουμε μια σειρά κριτηρίων όμως, ώστε η πλατφόρμα ΕΦΕ να μην είναι μόνο ε, μια καταγραφή φεστιβάλ, να μην είναι μόνο μια προκήρυξη ώστε να υποβάλουν αιτήσει στα φεστιβάλ και να συμμετέχουν σε ένα κατάλογο υποψηφίων φεστιβάλ. Ε, πρόκειται εδώ για μια πλήρη διαδικασία αξιολόγησης ποιότητας μέσα από τις αιτήσει ε, των φεστιβάλ online ε, που εξετάζονται σε διάφορα επίπεδα, σε διάφορες φάσεις από το τοπικό επίπεδο μέχρι το επίπεδο της Διεθνούς Κριτικής Επιτροπής. Τώρα, ε, αυτή η λατρεία των διασημοτήτων ε, μέσα από τα σήματα και τα βραβεία ε, και είπατε ότι πρέπει αυτό να το αποφύγουμε, δηλαδή να μην δώσουμε έμφαση στις διασημότητες. Όχι, αυτά που σας είπα για τα σήματα και τα βραβεία ε, δεν ε, είναι τα, χαρακτηριστικά της διαδικασίας μας αποτελούν ένα κομμάτι μόνο. Ε, γιατί ήμερο μπορεί οι οργανωτές φεστιβάλ να συναντώνται, να συζητούν για τα φεστιβάλ, τις δυνατότητες που έχουν και τις online δυνατότητες πάνω απ' όλα. Γιατί αν δημιουργήσουμε μια κοινότητα φεστιβάλ, 800-900 φεστιβάλ, στην πρώτη προσπάθεια για να υπάρχει το σήμα, αυτό θα είναι ένα δίκτυο όχι φίλων που γνωρίζει ο ένας τον άλλον, αλλά ένα δίκτυο οργανώσεων ε, που λειτουργούν κυρίως online και ε, λειτουργούν πάνω στη βάση των πληροφοριών και της γνώσης που έχουμε πλέον αποκτήσει για τα φεστιβάλ. Έτσι μπορούμε να, να εξασφαλίσουμε πρόσβαση για σε όλες τις πληροφορίες που έχουμε συλλέξει και που αφορούν το φεστιβάλ. Γιατί ένας Ολλανδός διοργανωτής φεστιβάλ δεν ξέρει τα τεκτενόμενα στη Γερμανία. Πολλές φορές μπορεί και κάποιοι Γερμανοί πολίτες να μην ξέρουν ή ενδιαφερόμενοι να μην ξέρουν ε, τα διάφορα είδη φεστιβάλ, δηλαδή τι γίνεται με τα φεστιβάλ μουσικής ή χορού, γιατί υπάρχουν διαχωρισμοί, είναι χωριστά όλα αυτά. Έτσι λοιπόν και σε εθνικό επίπεδο ε, υπάρχει δυνατότητα απόκτησης εποπτείας γενικότερης του χώρου, του τοπίου των φεστιβάλ και οι εθνικές αρχές μπορούν έτσι πιο εύκολα να σκεφτούν να δημιουργήσουν μια εθνική αρχή αρμόδια για τα φεστιβάλ που δεν υπάρχει σε όλες τις χώρες. Υπάρχει μια τέτοια αρχή μόνο σε κάποιες χώρες, όχι σε όλες. Τώρα για το πιλωτικό πρόγραμμα και την περιορισμένη εντολή του. όπω είπε και ο κύριος Κάρελ Πάλτακ προηγουμένω, εμείς φιλοδοξούμε το πιλωτικό αυτό πρόγραμμα να γίνει ένα πρόγραμμα ευρύτερο που πρέπει να γίνει ούτω ώστε να δημιουργήσουμε ένα σήμα και εκεί θα απευθύνονται όλα τα φεστιβάλ. Αυτό χρειάζεται χρόνο. Και αυτό είναι ένα μια πρόκληση, όχι πρόβλημα, πρόκληση που αντιμετωπίσαμε. Να φτάσουμε στα φεστιβάλ, να απευθυνθούμε επιτυχώς αυτά και να τα πείσουμε ότι αξίζει να μας χρησιμοποιήσουν γιατί ακόμα το σήμα δεν υπάρχουν. Δεν μπορούμε δηλαδή να τους ε, δώσουμε άμεση ε, ανταπόδοση βάζοντα το σήμα. Και βεβαίω τα φεστιβάλ ε, πολλές φορές δεν εντάσσονται σε ένα ευρωπαϊκό project γιατί λένε έχω απογοητευτεί τόσο πολύ από τη διαδικασία ολοκλήρωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν θέλω να το κάνω. Οπότε είχαμε μια ευκαιρία τώρα να αρχίσουμε ένα διάλογο και να ε, πείσουμε με τους οργανωτές φεστιβάλ ότι χρειάζεται ένα δίκτυο που θα εντάξει σε αυτό το διάλογο για την Ευρώπη τα φεστιβάλ. Και μια άλλη πρόκληση σε αυτό το επίπεδο είναι το οργανωτικό επίπεδο. Εμείς θέλουμε να αποκεντρώσουμε τη διαδικασία αυτή και να κάνουμε οργάνωση από κάτω προς τα πάνω. Από την άλλη βέβαια υπάρχει ανάγκη οργάνωσης ε, για ποιότητα. Μπορεί να υπάρχουν τα διάφορα κέντρα στις χώρες. Ε, τα κέντρα αυτά θα πρέπει να εφαρμόζουν τα κριτήρια και να παρακολουθούν τους εμπειρογνώμονες. Αυτό είναι μια πρόκληση γιατί είναι, υπάρχει ποικιλομορφία στην Ευρώπη. Στη Σουηδία γίνονται αλλιώ τα πράγματα από ό,τι στη Γερμανία ή στην Ουγγαρία. Και έτσι πρέπει να κάνουμε αποκέντρωση και από την άλλη να έχουμε ένα ποιοτικό ε, σημείο, ε, ε, πρότυπο αξιολόγησης, ένα κριτήριο αναφοράς, το οποίο θα ισχύει για όλους. Θα πρέπει δηλαδή να διασφαλίσουμε ορισμένα πρότυπα με αυτόν τον τρόπο. Σε επίπεδο πιλωτικού προγράμματο ελπίζουμε ότι θα συνεχιστεί η χρηματοδότηση γιατί πιστεύουμε ότι αυτό το πρόγραμμα θα πρέπει να παγιωθεί να εγκαθιδρυθεί στο πλαίσιο των ε, δραστηριοτήτων των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων. Δεν είναι μια πρωτοβουλία άπαξ, αλλά κάτι το συνεχές. Ελπίζομαι βέβαια ότι το Κοινοβούλιο θα παίξει το ρόλο του και θα κάνει τη δουλειά που πρέπει σε αυτή την Επιτροπή Πολιτισμού, ούτω ώστε να βρει τρόπο συνέχισης της χρηματοδότησης είτε του πιλωτικού προγράμματος ή γίνει μια προπαρασκευαστική ε, δράση ε, ως επόμενο βήμα. Αυτά είχα να σας πω, βέβαια δεν αναφέρθηκα σε κάθε ρωτώντα χωριστά, ε, μίλησα όμως ε, για την ποιότητα, το, τους ορισμούς, ε, τα κριτήρια και τη συνεργασία μας που ήδη έχει αρχίσει, μίλησα για τις προκλήσεις και τη σημασία συνέχιση που έχει να συνεχιστεί το πρόγραμμα αυτό σε επίπεδο ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ. Ήταν ε, περιστατωμένε οι απαντήσει σα, νομίζω. Πιστεύω ότι μπορούμε να εξετάσουμε την προοπτική. Νομίζω και η ε, Κομισιόν έχει εκφράσει θετική άποψη και το Κοινοβούλιο μπορεί να εξετάσει τη δυνατότητα για μια προπαρασκευαστική δράση ή για κάποια μορφή να καταστεί αυτή η εργασία και αυτή η πλατφόρμα κάτι που με τον καιρό θα <coughs> οικοδομηθεί, θα αναπτυχθεί με κάθε προσοχή σε όλες αυτές τις δυναμικές που φυσικά θα πρέπει να τις σεβαστούμε διαφορά, πολιτιστική διαφορά και ιδιαιτερότητες των διαφόρων φεστιβάλ. Νομίζω πως είναι πολλά υποσχόμενο αυτό το σχέδιο και ότι ανταποκρίνεται σε λίγο σε αυτή τη δυσκολία που αναφέρατε στην αρχή γιατί η γραμμή για την δημιουργική Ευρώπη ήταν, είχε πολλές δυσκολίες σε σχέση με το πόσα αιτήματα και πόσες δυνατότητες απάντησης γιατί το θέμα δεν είναι να δώσουμε μόνο οικονομική στήριξη αλλά να δώσουμε και ευκαιρίες, γνώσεις, δικτύωση, να διευρυθεί δηλαδή το κοινό και να προσφερθούν αυτές οι δυνατότητες και για αυτό το θέμα που μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρον για την Κομισιόν, για το... Την κινητικότητα δηλαδή των καλλιτεχνών είναι θέμα το οποίο μας είναι ιδιαίτερα προσφυλές γιατί είναι ένα από τα μεγάλα ζητήματα που έχουμε στην Ευρώπη. Σας ευχαριστώ όλους, ευχαριστώ όλους τους παρόντες από την ε, Ένωση. Ήταν ενδιαφέρουσα η δελεγή απόψεων και το ενδιαφέρον των συναδέλφων ήταν προφανές. Σας ευχαριστώ και πάλι, καλή δουλειά και έτσι κλείνουμε την ε, συνεδρίασή μας. Να ειδοποιήσω μόνο πω η επόμενη συνεδρίαση προβλέπει τι 4 και 5 Μαου, 4 Μαου στι 3 και τι 5 Μαου στι 9. Χωρίς μικρόφωνο η πρόεδρος. Επίσης να σας ενημερώσω ότι ίσως να κάνουμε μια έκτακτη συνεδρίαση στο Στρασβούργο γιατί ζητήσαμε την επαφή με τον Αντιπρόεδρο Άνσιπ. Τώρα θα γίνει η συνεδρίαση των συντονιστών. Θα συζητήσουμε τώρα το θέμα με τους συντονιστές γιατί είναι σημαντικό να γίνει η συνεδρίαση με τον Αντιπρόεδρο Άνσιπ πριν από την ανακοίνωση του σχεδίου για την ε, ε, ενιαία και αγορά. Σας ευχαριστώ πολύ και τώρα έχουμε τη συνεδρίαση των συντονιστών μας και παρακαλώ όσους δεν είναι συντονιστές να εγκαταλείψουν την αίθουσα. Ευχαριστώ.